ενέργειας, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και να σας πω κάτι στα ουγγρικά, στο τέλος, ότι έχουμε μία πρόταση ψηφίσματος που θα κλείσει τη συζήτηση, κλείνει τη συζήτηση. Και όντως την κλείνω, η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι την Πέμπτη. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας νύχτα.